Εντάξει, θα ήθελα να κάνω μια ανακοίνωση, ωστόσο. Έλαβα έτοιμα από την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών για τον κύριο Φεραντίνο που θα αντικαταστήσει τον Ούντο Μπούλμαν ως μέλος της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων. Ενστάσεις, όχι. Σας ευχαριστώ. Εγκρίνεται λοιπόν.